Κυρίε και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στο τελευταίο μας σημείο για σήμερα. Παρακαλώ τον εκλεκτό συνάδελφο, κύριο Μπουτικόφερ, να ολοκληρώσει τις ε, συνομιλίες του για το μέλλον της Ευρώπης και ιδίω για τι σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση-Σαουδική Αραβία. Ευχαριστώ. Ένα θερμό λοιπόν καλωσόρισμα στην μεγαλύτερά του Αντέλ Αλζουμπιέρ, τον ε, πρόεδρο τη Δημοκρατία τη Σαουδική ε, Αραβία, συγγνώμη, υπουργό εξωτερικών της ε, Σαουδική Αραβία. Σας καλωσορίζουμε στην Επιτροπή μας για να μιλήσουμε για την κατάσταση στη χώρα σας και την περιοχή του, κόλφου, του κόλπου. Ε, ανυπομονούμε να ακούσουμε για την άποψή σας για τις εξελίξεις, γιατί παρακολουθούμε την επίταση των σχέσεων και την αύξηση της έντασης μεταξύ ΙΠΑ ΕΕ και Ιράν. Ελπίζουμε ότι η αποκλιμάκωση, που είναι μια πήγουσα ανάγκη, θα γίνει πραγματικότητα. Θέλουμε να ακούσουμε τις απόψεις για τις σχέσεις σας με το Κατάρ, και ελπίζουμε ότι σύντομα το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου θα βρει μια λύση στην κρίση και για να δημιουργηθεί ξανά ε, μια κατάσταση σταθεροποίησης και εμπιστοσύνη στην περιοχή. Ακόμη και για την κατάσταση στην Ιεμένη, τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο αυτή τη στιγμή και δεν φαίνεται να υπάρχουν ε, ε, προοπτικές επίλυσης τώρα άμεσα. Ποιες είναι οι δικές σας απόψεις για τις προοπτικές αυτή την ε, πολύ ε, τραγική σύγκρουση. Επίση, θα θέλαμε να παρακολουθήσουμε το τι γίνεται με ένα blogger τώρα, Ιφ Μπαντάουι, ο οποίο κέρδισε το βραβείο Ζαχάροφ το 2015 για την ελευθερία τη έκφραση και ξεκίνησε για τέταρτη φορά απεργία πείνα το Σεπτέμβριο του 2019. Θέλουμε να επαναλάβουμε τη σημασία τη ε, παροχή βασιλική ε, χάρη υπέρ του. Χάριτος, υπέρ του. Ε, ευχαριστώ. Είναι χαρά μου να είμαι και πάλι εδώ και χαίρομαι που θα μπορέσουμε να συνομιλήσουμε. Ξέρω ότι έχετε περιορισμένο χρόνο, θα προσπαθήσω να συντομεύσω τα σχόλια μου. Λοιπόν. Η περιοχή μας είναι ενδιαφέρουσα και γεμάτη προκλήσεις. Μια σημαντική πρόκληση. Ε, είναι πολλά τα κράτη που συνεπάρχουν στην περιοχή Έχουμε τρομερούς φυσικούς πόρους, τρομερές δυνατότητες και πολλές προκλήσεις. Η Εμένη, Ισραήλ, Παλαιστίνη, Λιβάνο, Συρία, οι δραστηριότητες του Ιράν, το Ιράκ, το κέρας της Αφρικής, η Ερυθρά Θάλασσα, η χώρα του Σαχέλ, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, η Ινδία, Πακιστάν, δεν περνάμε ούτε μια στιγμή ανίας. Το 2020 θα πρέπει να δούμε όλες αυτές τις προκλήσεις μαζί για να προσπαθήσουμε να παρακολουθήσουμε σωστά τις εξελίξεις. Το σημαντικότερο είναι ο κόσμος. Ο κόσμος θέλουμε να βελτιώσουμε το βιωτικό του επίπεδο, ε, τη χώρα μας να την διατηρήσουμε προστατευμένη και να εφαρμόσουμε την ατζέντα μας για το 2030 να ανοίξουν νέοι τομεί για επενδύσει, να βοηθήσουμε την νεολαία και τι γυναίκε μα, να υπάρξει καινοτομία, εισρωή τεχνολογικών ε, εξελίξεων και λύσεων για, τον, για του πολίτε μα. Θέλουμε να είμαστε στην αιχμή των ε, εξελίξεων. Είμαστε μια χώρα με μετριοπάθεια, ε, ανεξιθρησκεία και ανεκτικότητα. Να δοθούν ευκαιρίε στου νέου μα εκ των οποίων 70% 70% των πολιτών μας είναι νέοι, κάτω των 30 και χρειάζονται ευκαιρίες, ευκαιρίες για να μπορέσουν να αριστεύσουν. Και η Σαουδική Αραβία να γίνει πλουσιότερη, ε, καλύτερη και δυνατότερη. Χρειαζόμαστε βαθιές κοινωνικές αλλαγές, αυτό είναι ο στόχος μας για το 2030 και πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε αυτούς τους τομείς που προανέφερα, ιδίως ό,τι αφορά το δικαίωμα του συναθρίζεστε σε δημόσιου χώρου, την ψυχαγωγία, την, τα δικαιώματα των γυναικών και την άσκησή του. Οι γυναίκε οδηγούν πλέον, μπορούν να ταξιδεύουν χωρί την άδεια κανενό, όπω οι άντρε. Έχουν πρόσβαση σε όλε τι θέσει εργασία στο δημόσιο τομέα. Μπορούν να παίρνουν ίδιους μισθούς για με, ίδια δουλειά με τους άντρες, για περιβαλλοντικά ζητήματα, ε, απασχολούνται επίσης και ταυτόχρονα μεταρρυθμίζουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Κοιτάζουμε να ε, εξαλείψουμε τις εξτρεμιστικές τάσεις και να προάγουμε την μετριοπάθεια. Όποιο κοιτάξει σήμερα τη Σαουδική Αραβία θα δει μια μετριοπαθή, ανεκτική, σύγχρονη, ε, κοινωνία. Με σφάλματα, σίγουρα αναπόφευκτα, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση στο βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας. Ήδη έχουμε αρχίσει να βλέπουμε αυτά τα αποτελέσματα. Έχουμε δει μια σχετική αύξηση στις ξένες επενδύσεις στη Σαουδική Αραβία πέρσι. Τεράστια αύξηση στον αριθμό επιχειρηματιών που άνοιξαν εταιρείε στη Σαουδική Αραβία Κάτι που είναι ένα πολύ θετικό δείγμα για το ότι δείχνουν εμπιστοσύνη στη σαουδαραβική οικονομία και τις διαδικασίες μεταρρύθμισης μας, καθώς και το μέλλον της χώρας. Ξέχασα να αναφέρω ένα στατιστικό στοιχείο. Βάσει ενό Υπουργείου, του Υπουργείου Εσωτερικών και Επενδύσεων, το 39% των επιχειρηματιών στην Σαουδική Ραβία σήμερα είναι γυναίκε. Αυτό είναι τεράστιο, τεράσ, τεράστια σημασία μάλλον το 39% των φοιτητών σε πανεπιστημιακή κολέγια είναι γυναίκες. θα συνεχίσουμε λοιπόν σε αυτή την πορεία γιατί είναι προ όφελο τη ίδια τη κοινωνία τη Σαουδική Αραβία. Ε, σε ό,τι αφορά το Κατάρ που αναφέρατε. Έχουμε προβλήματα με το πώ το Κατάρ στηρίζει την τρομοκρατία και τον εξτρεμισμό. Υπάρχει χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων όπως Χεσμολά στο Ιράκ και άλλοι ε, και με λίτρα που πληρώνονται σε εκπροσώπους των ε, οργανώσεων αυτών. Έχουμε θέματα με το Κατάρ και την ανάμειξη στις ιστορικές μας προθέσεις. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα αλλάξει η στάση τους και θα αρχίσουν να συμπεριφέρονται σαν μια πειθαρχημένη χώρα. Έχουμε προβλήματα με τις πλατφόρμες μέσων ε, μαζικής ενημέρωσης και με άτομα παρότρινσης σε μίσος. Προσπαθούμε να τα εξαλείψουμε αυτά. Τα προβλήματα υφίστανται. Οι φίλοι μας από το Κατάρ εξαρτάται αν θα αλλάξουν τη συμπεριφορά τους και τις τάσεις τους για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Κοιτάξαμε να βεβαιωθούμε ότι στα πλαίσια του Συμβουλίου Συνεργασίας του των χωρών του Κόλπου και στο επίπεδο υπουργικών συνόδων δεν υπάρχουν ε, δυσκολίες συνάντηση, η στρατηγική εκπαίδευση δεν επηρεάζεται από αυτή την κρίση. Θέλουμε να παραμείνει η ενότητα των χωρών ε, του κόλπου και τη συνεργασίας τους. Και αυτή η κρίση να επιληθεί. Με ρωτήσατε για τον ε, Ραΐφ Μπεντάουι. Το δικαστικό σύστημα όμω είναι ε, ανεξάρτητο όπω στι χώρε σα. Είναι δική του απόφαση των δικαστών το τι θα γίνει. Και νομίζω ότι θα πάψω εδώ. Θα σταματήσω γιατί δεν θέλω να μονοπολίσω τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Αλζουμπία. Και πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους, να καλωσορίσω και τον πρέσβη από το Βασίλειο τη Σαουδική Αραβία, τακτικό επισκέπτη του Ευρωκοινοβουλίου. Συνάδελφοι, έχουμε μισή ώρα στη διάθεσή μα για να έχουμε διάλογο με τον αποστεκλημένο μα από τη Σαουδική Αραβία. Παρακαλώ, ζητήστε το λόγο, όπω ήθιστε. Ξεκινάμε με τον κύριο. Βετλίγκα. Α, όχι, ο κύριος Γκάλαγαρ πρώτα. Καλώς. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ, στην Επιτροπή μας αυτή. Σας ευχαριστώ για τις εξηγήσεις που μας δώσατε για τους στόχους σας στο εσωτερικό. Άκουσα για μετριοπάθεια, για ανοχή. Χαίρομαι για αυτά. Και κυρίως όταν πρόκειται για τα δικαιώματα ε, της γυναίκας, το οποίο αναφερθήκατε. Εύχομαι αυτό το πνεύμα μετριοπάθειας και ανοχής να εξαχθεί και εκεί που χρηματοδοτεί η Σαουδική Αραβία τζαμιά, είτε πρόκειται για την Τινησία, είτε πρόκειται για τους Λαμαμπάτ, ο κόσμος ο, μου λέει ότι η Σαουδική Αραβία χρηματοδοτεί. Και από ό,τι φαίνεται πρόκειται για την σαλαφιστική εκδοχή, την πιο σκληρή. Αν λοιπόν έχετε στόχους μετριοπάθειας και ανοχής, σας παρακαλώ να φροντίσετε αυτές οι αρχές να ε, φτάσουν και εκεί όπου χρηματοδοτείτε. Τώρα η ερώτησή μου δεν έχει να κάνει με το άμεσο μέλλον και τις σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία και τις γειτονικές χώρες, αλλά για πιο μακροπρόθεσμα. Θα συμφωνούσατε να έχετε κάτι σαν και αυτό που είχαμε και εμείς πριν από 40 χρόνια μια διάσκεψη για την ασφάλεια και την ανάπτυξη ή τη συνεργασία στην περιοχή σας, όπου να συμμετέχουν όλες οι ενδιαφερόμενες χώρες και άρα να είσαστε υποχρεωμένοι όλοι να καταλήξετε σε ένα κοινό και ειρηνικό μέλλον για όλους σας. Είναι μια προοπτική που θα βλέπατε χωρίς προϋποθέσεις. Ε, στο τέλος εμείς καταφέραμε κάτι θετικό. Ευχαριστούμε, Μιχαήλ Γκάλερ. Η Μαρία Ρένα τώρα, μέρους των Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ πολύ. Έχω κάποιες ερωτήσεις για το θέμα των δικαιωμάτων ε, του ανθρώπου. Το Φεβρουάριο του 2018 το Κοινοβούλιο μας ενέκρινε ψήφισμα ε, κατεπήγοντος και πρόκειτο για αυτούς που υποστηρίζουν τα δικαιώματα των γυναικών στη Σαουδική Αραβία και κυρίως τους αγωνιστές οι οποίοι κρατούνται χωρίς να τους έχει ε, αποδοθεί κατηγορία και από την άλλη υπάρχουν πάρα πολλέ επικρίσει σε βάρος της Σαουδική Αραβίας από αυτού. Τι θα γίνει με την απελευθέρωσή τους κυρίω, γιατί ακριβώς ε, θέλανε να προωθήσουν το δικαίωμα των γυναικών στην οδήγηση, κάτι το οποίο τελικά έγινε νόμος. Τι θα γίνει με τους αγωνιστές αυτούς, θα απελευθερωθούν. Δεύτερον, βραβείο Σαχάροφ. Ο κύριο Μπανταουή ο οποίος βραβεύτηκε το 2015, φυλακίστηκε το 2012, η κατάσταση υγείας του είναι ανησυχητική και θα θέλαμε να υπάρξει απόφαση απελευθέρωσής του για ιατρικούς λόγους. Μπορείτε να λάβετε υπόψη σας αυτό το αίτημα το οποίο εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να απελευθερωθεί ε, αυτός που τιμήθηκε με το βραβείο Ζαχάροφ. Έρχομαι τώρα σε πιο πολιτικά ζητήματα, για 400 εκατομμύρια γεμενίτες, 12 εκατομμύρια παιδιά εξαρτώνται από την ανθρωπιστική ε, βοήθεια. Ε, υπάρχει συμφωνία της Τοκόλμης που στηρίζουμε και η δέσμευση της Οδικής Αραβίας για να υπάρξει η ειρήνη στην περιοχή. Τέλος, για το Ιράν. Ποια είναι η στάση της Οδικής Αραβίας στην πρωτοβουλία για την αποκλιμάκωση Ε, στις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων, ε, Πολιτειών και Ιράν. Είναι Φανβίζε από το Ρινιού. Ευχαριστώ πολύ. Ε, με ξοχώτης. Και εγώ μιλάω εκ μέρου τη Υποπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αναγνωρίζουμε ότι έχει επιτευχθεί η πρόοδο στη Σουδική Αραβία, κυρίω όσον αφορά τα δικαιώματα τη γυναίκα ε, και ευχαριστούμε. Όμω, Υπάρχουν και 13 ακτιβίστριες οι οποίες από το 2018 έχουν συλληφθεί για τη δράση τους. Επρόκειτο για το δικαίωμα των γυναικών ε, στην ε, οδήγηση, για το δικαίωμα της υπηκότητας κτλ. Ξέρω ότι 5 από τις 13 παραμένουν στη φυλακή σήμερα. Νεκατζού, Σαρμαρβοντάβιν, Νασίμα Τσάντα, Νούφα και η Αλσαχράνη. Συχνά ακούμε ε, το άλοθη της ασφάλειας. Πώς όμως εξηγείται ότι κάποιες από αυτές ε, πήγαν στη φυλακή και τους αποδόθηκαν κατηγορίες, ενώ η διεθνή Αμνηστία μιλάει υπέρ τους. Έπειτα έχει ερευνήσει η κυβέρνηση τι, τα όσα έχουν ακουστεί για βασανισμούς σε βάρος τους και σε βάρος άλλων υποστηρικτών ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και φαίνεται ότι μία από αυτές νασίμα βρέθηκε στην απομόνωση από τις αρχές του 2019. Ευχαριστούμε. Από τους πράσινους κάποιος. Χάνα νόημα. Ναι. Ευχαριστώ. Όπως και άλλες δύο συνάδελφοι από την Υποπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, που είπαν πράγματα πολύ του The Point, έτσι και εγώ θέλω να θίξω κάποιες πτυχές για πιθανότητα και δυνατότητα συνεργασίας. Η επίσκεψή σας έρχεται σε μια καλή στιγμή. Υπάρχει κλιμάκωση μετά τη δολοφονία του Σουλημάνη. Η κατάσταση στην περιοχή μπορεί να επιδεινωθεί πολύ γρήγορα. Και είναι προς το συμφέρον όλων τέτοια κλιμάκωση να μην επαναληφθεί στο μέλλον. Αντίθετα, θα θέλαμε αποκλιμάκωση. Όμως οι συγκρίσεις, όπως και η δολοφονία του Σλεμανί, αλλά και οι επιθέσεις στα πετρέλαια της οδικής Αραβίας δεν βοηθούν. Και είπα το εκπρόσωπος που είχαμε πριν, η κυρία Μογκερόνη, ε, προσπάθησε να πετύχει μία διάσκεψη όπου να συμμετέχουν οι χώρες της περιοχής και το Ιράν και το Ιράκ και η Σαουδική Αραβία. Οπότε η ερώτησή μου είναι, εσείς πώς αξιολογείτε τη δυνατότητα να υπάρξει μια τέτοια περιφερειακή προσέγγιση. Είναι το θέμα της ελπίδας. Και έχω και άλλη μία ερώτηση. Άκουσα να μιλάτε για ένα σωρό πράγματα που θέλετε να κάνετε στη Σουδική Αραβία ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανθρώπινα δικαιώματα, λύση στην Ιεμένη, γυναίκες, ελευθερία έκφρασης. Πολύ καλός ο κατάλογος και έχουμε δει κάποια συγκεκριμένα βήματα. Όμως θα ήθελα να επιταχυνθεί κάπως η πορεία. Να δω εσείς τι μπορείτε να κάνετε για αυτά. Πώς θα μπορούσατε εσείς και σε Σαουδική βία να συνεργαστείτε για να επιταχυνθεί η πορεία. Είπατε, μια κοινωνία με μετριοπάθεια, ανοχή και τη συμμετοχή όλων. Πώς θα το καταφέρετε αυτό. Ευχαριστούμε. ECR. Νόιμαν. Εδώ. Μπροστά μας. Α, όχι. Είναι ο κύριος Φανόρδεν τώρα που κάθεται εδώ μπροστά μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε. Η μεγάλη απειλή στην περιοχή σας είναι το Ιράν βέβαια. Αλλά η άλλη μεγάλη δύναμη στην περιοχή είναι η Τουρκία βέβαια. Που είναι σύμμαχος κλειδί στο ΝΑΤΟ. Εσείς βλέπετε δυνατότητα βελτίωσης των σχέσεων Σαουδικής Αραβίας με την Τουρκία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Τζέφρι. Ο κύριος Κούλογλου από την ΚΟΕ. Ελληνικά θα μιλήσετε φαντάζομαι. Ε, ε, Να γιατί όχι, αν ε, καταλαβαίνει ελληνικά η αυτό Okay, let's go on with English. Ας συνεχίσουμε στα αγγλικά παρόλα αυτά. You, have said some very nice. Κύριε Υπουργέ, είπατε πολύ όμορφα λόγια, τα οποία απευθύνατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ταυτόχρονα μιλήσατε και για την ελευθερία έκφρασης, τα δικαιώματα των γυναικών. Όμως αυτή τη στιγμή υπάρχουν γυναίκες που έχουν φυλακιστεί γιατί αγωνίστηκαν για τα δικαιώματά τους. Έρχεστε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και υπάρχει κάποιος, ο κύριος Μπανταουή, που έχει τιμηθεί με το βραβείο Σαχάροφ το μεγαλύτερο ε, βραβείο για τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βρίσκεται ακόμα στη φυλακή. Κάτι δεν θα έπρεπε να μας έχετε πει και για αυτά. Στην Ιεμένη ξέρουμε ότι επικρατεί μια κατάσταση ανθρωπιστικής καταστροφής και η Σαουδική Αραβία φέρει ευθύνη για αυτή την καταστροφή και τη συμμετοχή της ε, στον εμφύλιο πόλεμο. Δεν είπατε τίποτα από αυτού. Και τέλος. στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας απασχολεί ιδιαίτερα το θέμα της δολοφονίας ε, του ε, δημοσιογράφου Κασόντζη. Η δίκη που τελικά έλαβε χώρα, στην ουσία τελικά απείλαξε την ηγεσία του βασιλείου, που για τους περισσότερους από εμά είναι απόλυτα υπεύθυνη για τη δολοφονία. Λυπάμαι αλλά κάτι πρέπει να μας πείτε. Και για αυτή την υπόθεση. Κάποιοι μυστικοί πράκτορες ε, καταδικάστηκαν, λες και δρούσαν αυτοβούλος. Ελπίζω εγώ και άλλοι συνάδελφοι που σας επέκριναν να μην καταλήξουμε ε, δολοφονημένοι και κατακριουργημένοι. Τέσσερις ακόμα ομιλητές. Πριν δώσουμε το λόγο στον ομιλητή, Λέγκε, Βαζέσκου, Χούβερτ και Αστροβίτσιους. David Ευχαριστώ. Παρά την ε, διαδικασία στη Σαουδική Αραβία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ και πολλοί Ευρωπαίοι ακόμα, έχουμε σημαντικές επιφυλάξεις ό,τι αφορά τη συνεχιζόμενη χρήση του μέσου της κράτησης ως πολιτικού μέσου. Ε, υπάρχουν ανώτερα μέλη ε, της βασιλικής οικογένειας, όπως ο Μπιν Αμπτούλα, που κρατούνται χωρίς δίκη ενώ υπάρχουν δημοσιογράφοι, blogger που ε, έχουν ε, μπει στη φυλακή για χρόνια επειδή εξέφρασαν ε, τη γνώμη τους και μόνο, όπως είναι και το δικαίωμά τους. Ποια θα είναι η διαδικασία για την απελευθέρωσή τους, εφόσον πρόκειται για θεμέλιο λίθο του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Βαζέσκου. Ευχαριστώ. Καλώς ήλθατε κύριε Υπουργέ. είναι περίπλοκο το ερώτημα, αλλά μπορεί να καταφέρετε να απαντήσετε. Υπάρχει μια τρομερή ε, σύγκρουση αυτή τη στιγμή στην ε, περιοχή για το ποιος θα κυριαρχήσει μεταξύ Ιράν και Σαουδικής Αραβίας. Τελικά, ποια είναι τα ωφέλη για τους ε, Σαουδάραβες, για το λαό σας, εάν εσείς και το Ιράν βρίσκεστε ε, στο διγυναικέ αυτή την, ε, σε αυτόν τον ανταγωνισμό για να κυριαρχήσετε στην περιοχή. Ευχαριστώ, Μάρτιν Χάουαρντ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, Αυτοξοχώτης, Αλέκουμ. Κάθε φορά που σας έχω ε, συναντήσει, με έχετε υποδεχθεί με πολύ ευγένεια. Καλώς ήρθατε λοιπόν και από πλευρά μου. Δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι ε, στη Σαουδική Αραβία υπάρχουν ε, κατάφορες παραβιάσεις ανθρωπινών δικαιωμάτων κατά ε, ακτιβιστών και διανοωμένων που απλώς εξέφρασαν τις απόψεις τους δημοσίως ή κατηδίαν. 194 ε, άνθρωποι εκτελέστηκαν στα Δική Αραβία πέρσι, αριθμός ρεκόρ, 37 άτομα σε μία και μόνο ημέρα τον Απρίλιο. 90 άλλο θα πει, για τους οποίους υπάρχουν σημαντικές ε, πηγές προβληματισμού, τρία παιδιά και υπάρχουν πολλές κατηγορίες ε, για βασανιστήρια ή έλλειψη δίκαιης δίκης. Και συνάδελφός μου η Ρίνα, ήδη ανέφερε τον Χουσένο Ασλούβ, Χασίνα Σάντα και άλλες γυναίκες που έχουν φυλακιστεί για υποτιθέμενα δικήματα που στις χώρες μας ε, απλά δεν θα σημαίναν τίποτα. Θα, θα περνούσαν απαρατήρητες αυτές οι ενέργειες. Και από την άλλη έχουμε και τον Αϊφ ε, Αμπατάουι που μένει στη φυλακή επειδή ξεκίνησε το λεγόμενο ε, σαουδαραβικό ε, δίκτυο, φιλελεύθερο δίκτυο που δεν είναι και κάτι που ακούγεται τόσο απειλητικό θέλετε να βλέπουμε τη Σαουδική Αραβία ως ε, μία μετριοπαθή, σύγχρονη, ε, συμπεριληπτική κοινωνία. Αλλά δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε να σας δούμε έτσι. Έω ότου επιτέλου, αντιμετωπίσετε αυτέ τι κατάφορε παρεμβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, έχετε εξαιρετικά αρνητική εικόνα στην διεθνή κοινότητα και αν θέλετε να σα βλέπουμε ω φίλου, θα πρέπει αυτό να αλλάξει. Ο κύριος Στραβίτσιος. ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, καλώ ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χαιρετίζουμε πολλού και υποδεχόμαστε πολλού προσκεκλημένου, στου οποίου μιλούμε με κάθε ειλικρίνεια και αυτό θα κάνουμε και μαζί σα. Είναι πολλά υποσχόμενη η παρέμβασή σα και εύχομαι η χώρα σα ε, να αλλάξει ε, προς το καλύτερο, προς περισσότερη ε, ανοχή και σεβασμό των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Από τότε όμως, ε, εφόσον μάλλον ο Ανρί Μπαντάουι παρότι έχει τιμηθεί με τον Ρίο Σαχάροφ, μένει στη φυλακή ενώ περιμένει την, ε, ε, να δικαστεί. Εμείς αναγκαζόμαστε να ζητήσουμε την ανεφόρον απελευθέρωσή του. Δεν μπορούμε να σιωπήσουμε ως προς αυτό. Πρέπει να τον δούμε ελεύθερο και σώκια βλαβή, ακόμα και στα δική Αραβία. Δεύτερον, θα ήθελα πραγματικά να ακούσω ένα σχόλιο για τη δίκη στην υπόθεση Κασότζη, ο οποίος δολοφονήθηκε βάναυσα και μάλιστα στην επικράτεια της ε, ε, Πρεσβείας. Πέραν ε, της, ε, του ομού χαρακτήρα της ε, δολοφονίας σας, πρέπει εσείς να σχολιάσετε. Ελπίζω να συμφωνείτε. Ω Δημοκρατική Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσβλέπει ε, στη συνέχιση τη συνεργασία με, με τη Σαουδική Αραβία. Αλλά το μπαλάκι έχει περάσει στο δικό σα γήπεδο. Ελπίζω να το κατανοείτε κι εσεί. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ για τι τόσο απεθ... άμεσε και ειλικρινεί έντιμε ερωτήσει σα. Κύριε Υπουργέ, μπορείτε να απαντήσετε με όποια σειρά θέλετε. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω από την Ιεμένη και την κρίση εκεί. Στην οι θέλαμε να περάσουμε σε μια μετάβαση τον πρόεδρο Σάιλ σε κάτι καινούριο. Όμως απήχθησαν άνθρωποι και ε, ξαφνικά υπήρχε ένα καθεστώς τρομοκρατία και βίας. Όταν ένας από τους αντιπολιτευόμενους ε, προσπάθησε να κάνει κάτι, τον ε, κυνήγησαν, τον φυλάκισαν, ζήτησε βοήθεια εννιά μήνες μετά. Πιέσαμε για κάθε πολιτική λύση. Και για απελευθέρωση των 70 κρατουμένων έχουμε τις, ε, τους βαλιστικούς πυράβλους των Χούθη που προσπαθούν να βάλουν κατά τις χώρες μας, οδηγούν τον κόσμο σε ε, λοιμό ο συνασπισμό και η συμμαχία μα προσπαθεί να εξηγήσει γιατί είναι υπεύθυνοι οι Χούθη για όσα συμβαίνουν. Έχουμε δώσει 40 ε, εκατομμύρια δολάρια μέχρι τώρα ω ανθρωπιστική βοήθεια στην Ιεμένη και οι Χούθη εμποδίζουν την ε, προσέλευση τη ανθρωπιστική βοήθεια. Κανεί δεν λέει τίποτα για τα θέματα αυτά στο σώμα σα, οι Χούθη. Έχουν ε, θέσει εκατομμύρια ανάρκε έχουν κοστίσει τη ζωή των ε, κατοίκων τη Εμένη και δεν λέει κανεί τίποτα. Εμεί τα γνωρίζουμε όμω και κάτι δεν πάει καλά με την εικόνα που παρουσιάζεται. Εμεί πιέζουμε με τον Μάρτιν Γκρίφιθ προκειμένου να κινηθούμε σε μια πολιτική λύση στην Εμένη. Έχουμε εργαστεί σκληρά για την αποκλιμάκωση. Οι Χούθοι όμω περιόρισαν μόνο τι βαλιστικέ του επιθέσει κατά τη Σαουδική Αραβία και έχουν περιοριστεί κάπω οι επιχειρήσει στο έδαφο τη Εμένη σε όσα έχουν σχέση με τα αεροδρόμια και τους λιμένες ή την αντιλαγή κρατουμένων υπάρχει κάποια σχετική πρόοδος, αλλά δεν έχουμε ακόμα μια σαφή πολιτική λύση. Η ιδέα ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τον πόλεμο στην Εμένη δεν ισχύει. Η Χούθη είναι η αυτουργιακίνη ε, είναι υπεύθυνη για τις φρικαλαιότητες, όχι εμείς και ο κόσμος τι να το ξεχνάει. Κάτι άλλο που συζητήσαμε ήταν το Ιράν. Η Σύνοδο Συμφιλίωση Από το 1979 δεν έχουμε δει τίποτα άλλο παρά καταστροφή από το Ιράν. Έχουμε απλώσει το χέρι μα ε, χείρα φιλία και δεν βλέπουμε καμία απάντηση. Έχουν δολοφονήσει οι μα. Έχουν, ε, επανειλημμένω έχουν ε, επιτεθεί κατά τη πρεσβείες μα στο Ιράν. Έχουν βομβαρδίσει εγκαταστάσει στη Σαουδική Αραβία. Έχουν προσπαθήσει να αποσταθεροποιήσουν τον Μπαχρέν και το Κουβέιτ την Ιεμένη έχουν προσπαθήσει να δημιουργήσουν αντίπαλες φρατρίες και πιστεύουν ότι η αρχή της εξαγωγής της επανάστασης είναι το παν. Δεν πιστεύουν στην κυριαρχία, την εθνική κυριαρχία των εθνών. Πιστεύουν ότι το... οι ΣΥΤΕΣ είναι δικοί τους και είναι λες και να λένε οι Ιταλοί ότι όποιος είναι καθολικός είναι μόνο Ιταλός. Δεν πάει έτσι. Δεν πιστεύουμε. Εμείς πιστεύουμε στην αρχή της μη παρέμβασης. Δεν θέλουμε εξάπλωση τη τρομοκρατία στον κόσμο. Γι' αυτό έχουμε πρόβλημα με το Ιράν. Γι' αυτό μα ενοχλεί. Εάν οι Ιρανοί άλλαζαν συμπεριφορά, θα είχαμε και κάποια δυνατότητα συνεννόηση. Αλλά αν δεν το κάνουν, τι να κάνουμε και τι να επιδιώκουμε. Από το 79 δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν μα έχει πάει πουθενά οποιαδήποτε κίνηση. Είχαμε πρόσφατα διαδηλώσει στο Ιράν. Είχαμε και Σιήτες που διαμαρτύρονται στο Ιράν κατά τις ε, σε εμά κατά τις επιρροές του Ιράν. Και υπήρξαν μόνο ε, βομβαρδισμοί των εγκαταστάσεών μα. Αυτή είναι η απάντηση του Ιράν για όσο συμβαίνει στην περιοχή. Η πίεση λοιπόν πρέπει να συνεχιστεί και στο Ιράν και προκειμένου το Ιράν να αλλάξει συμπεριφορά και στάση και να τηρήσει τους κανόνες του διεθνούς δικαίου που ορίστηκαν μετά τη συνθήκη της Βεσφαλίας. Είναι εύκολο να κάθεται κανεί στι Βρυξέλλε και να λέει γιατί δεν κάθετε να συζητήσετε. Ε, γιατί δεν σα έρχονται βροχή πύραυλοι εδώ πέρα. Ούτε δολοφονούνται οι εκπροσωποί σα, ούτε οι πρεσβείε σα ε, δέχονται βομβιστικέ επιθέσει. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε με το Ιράν και αυτό είναι και το πρόβλημα που έχει ο κόσμο με το Ιράν. Έχουμε το θέμα του Συμβουλίου Συνεργασία των Χωρών του Κόλπου. Έχουμε το θέμα τη ε, χρηματοδότηση τη Δημοκρατία, κάτι πρέπει να πάψει τον... και πρέπει να αποφασίσουν οι Ιρανοί εάν θέλουν επανάσταση, ε, εάν μπορεί να συνεχιστεί αμύωτη η δράση τους και αν θέλουν να είναι ένα κανονικό κράτος πρέπει να συμπεριφερθούν αναλόγως για να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε συζήτηση μεταξύ τους Αυτά για τα θέματα του Ιράν. Τώρα για τον εξτρεμισμό και την εξαγωγή του εξτρεμισμού. Το Αφγανιστάν είχαμε, και στα Βαλκάνια, είχαμε οργανώσεις που δρούσαν δίθεν φιλανθρωπικά και ανακαλύψαμε ότι είναι εξτρεμιστικές. Ε, το ανακαλύψαμε και τις εξαρθρώσαμε τις, τις οργανώσεις αυτές. Ε, το ανακαλύψαμε εντό και εκτό Σαουδική Αραβία για τη χρηματοδότηση τη τρομοκρατία. Μόλι βρούμε κάποιον που κάνει κάτι τέτοιο, τον τιμωρούμε. Δεν έχει σημασία που ε, δείχνει κανείς και εκδηλώνει την έλλειψη ανεκτικότητας και το μίσος, πάντοτε γυρνάει μπούμεραν αυτό. Οπότε οι εξτρεμιστές δεν είναι οι Βρυξέλλες, είναι η Μέκα και είναι το κέντρο του Ισλάμ, υποτίθεται. Εμείς όμως να είμαστε συγκαταβατικοί ως προς τους ανθρώπους που χρηματοδοτούν την τρομοκρατία για τον εξτρεμισμό, είναι εντελώς παράλογο να θεωρείτε ότι μπορεί να συμβαίνει συνεργαζόμαστε με δυνάμεις παγκοσμίω για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα. Έχουμε πρόβλημα με την ε, μουσουλμανική αδερφότητα που έχει εξαπλωθεί παγκοσμίω, προσπαθεί να επηρεάσει κυβερνήσει, πιέζει και δημιουργεί εξτρεμιστικά φαινόμενα, αλλά δεν το έχουμε σχεδιάσει εμεί αυτό. Υπάρχουμε, μιλάμε για ζητήματα τα οποία είναι κατάλοιπα του παρελθόντο εδώ και τέσσερι εμείς είμαστε το βασικό θύμα και είμαστε και πρωταγωνιστές στον αγώνα κατά της δημοκρατίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δράσουμε σε επίπεδο καρδιάς και μυαλού και να καταπολεμήσουμε τον εξτρεμισμό. Ο ρόλος της Ευρώπης είναι σημαντικό στην περιοχή μας. Έχουμε ιστορικέ σχέσει, τεράστια οικονομική δύναμη μαζί, ε, πολιτική σύνεση. Κάθε τομέα στον οποίο αναφέρθηκα στην αρχή έχει, είναι ένας ε, χώρο που έχει να διαδραματίσει κάτι η Ευρώπη, η Συρία, το Ιράκ ή η εμενη Δεν μιλάω για οικονομική μόνο βοήθεια, αλλά και κυριολεκτικά. Ο κόσμος σας, οι άνθρωποι σας, ένοπλοι πολεμούν ε, τον Ταϊς στη Συρία και το Ιράκ. Γυναίκες και άνδρες πολεμούν για τη σταθερότητα ε, στο Αφγανιστάν. ή στις χώρες του Σαχέλ για την καταπολέμηση του Μπόκο Χαράμ για την καταπολέμηση της πειρατείας στον κόλπο του Άνταμ. Ε, πρέπει να υπάρξει συνεργασία λοιπόν. Χρειάζεται και στη σημαντική και την περιοχή μας. Τώρα για τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σας ανέφερα για τα περίπτωση του κυρίου Ραφάου και το Σαουδαραβικό δικαστικό σύστημα. Όμω δεν θέλουμε να δεχόμαστε κηρύγματα για το πώ θα πρέπει να λειτουργεί το δικαστικό μα σύστημα. Αν δούμε την πρόσφατη ιστορία, μερικά από τα φρικτότερα εγκλήματα έχουν λάβει χώρο σε αυτή την Ήπειρο. Από εδώ. Και οι συνέπειε των εγκλημάτων αυτών επέτρεψαν στι κοινωνίε σα να εξελιχθούν η δημοκρατία, το κράτο δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν ήρθαν μια ανοιχτή στην Ευρώπη. Οπότε πάψτε τα κηρύγματα, γιατί και εμεί κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έχουμε δικαστικό σύστημα, είναι ανεξάρτητο και δεν δεχόμαστε αμφισβητήσει για το πώ λειτουργεί. Είμαστε μια χώρα εθνικά κυρίαρχη. Ε, δεν είμαστε καμιά μπανανία. Οπότε θα πρέπει να σέβεστε τι αποφάσει του δικαστικού μα συστήματο. Σε ό,τι αφορά το Human Rights Watch και τι σχετικές καταγγελίες. Κάποια στιγμή η οργάνωση αυτή στη Σαουδική Αραβία είχε αμφιλεγόμενες ε, διαπιστώσεις. Μας είχαν κατηγορήσει ότι είχαμε επιτρέψει να εξαπλωθούν εκφράσεις μίσους. Τι ακριβώς όμως θέλετε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα αντίθετα ταυτόχρονα. Έχουμε συνεργαστεί με το Human Rights Watch, έχουν έρθει στη Σαουδική Αραβία επανειλημμένως, αλλά δεν τα λένε αυτά που διαπίστωσαν στη μελέτη τους. Τώρα το γεγονός ότι τρεις άνθρωποι καταδικάστηκαν σε θάνατο, και το αναφέρατε εδώ πέρα, διότι είχαν ε, διαπράξει εγκλήματες βάρος όταν ήταν έφηβοι ακόμα, δεν ε, επιβάλαμε θανατική ποινή σε κάποιον ε, όταν ήταν πριν τα 18 και έχουμε και μέγιστη διάρκεια κράτησης για 10 χρόνια όταν κάποιο είναι 118. Δεν επιβάλλουν θανατική καταδίκη σε κάποιον για κάτι που διαπράχθη πριν τα 18. Ε, προέκυψαν φήμες κάποια στιγμή για την Σαουδική Αραβία και ότι κάποιο καταδικάστηκε σε θάνατο όταν ήταν 15, ε, ε, από όταν ήταν 15 για κάτι που διέκαμπε τότε και θα καταδικαστεί μόλις γίνει 18. Μα είναι παράδεκτο και εδώ και στο σώμα σας και σε άλλα ε, κοινοβουλευτικά σώματα βάσει θυμών Δεν έχουν συμβεί τέτοια πράγματα. Είναι διαδόσεις. Κανένα τέτοιο νέος δεν καταδικάστηκε σε θάνατο, ούτε πρόκειται να θανατωθεί. Το έγκλημα που είχε διαπράξει ήταν ε, κάτι που διαπράχθηκε πριν την ηλικία των 18. Σε κάποιε περιπτώσει, στα 16 στα 17 έχουν διαπραχθεί εγκλήματα. Αλλά άλλα που τιμωρούνται με θανατική καταδίκη ε, διπράθησαν όταν ήταν 22. Καταδικάστηκαν για τα εγκλήματα μετά την ηλικία των 18. Όμως τα μέσα το προβάλλουν αλλιώς. Κάποιες από τις οργανώσεις αυτές όπως η Rights Watch, Human Rights Watch, αναφέρονται στα προηγούμενα εγκλήματα, τα προγενέστερα και λένε ότι για εκείνα καταδικάστηκαν. Όχι, δεν ισχύει. και για τις γυναίκες, τις κρατήσεις. Το θέμα του Τζαμάλ Κασότζη. Ήταν ένα σοβαρότατο σφάλμα. Θα πληρώνουμε το τίμημα για πάρα πολλά χρόνια από τη θεωρία. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είχαν το Abu Ghraib ε, οι εγκαταστάσεις ήταν υπό αμερικανικό έλεγχο. Διαπίστωσαν όμως κάτι στραβό. Όχι. Αυτό που έκαναν οι ΗΠΑ ήταν ότι ερεύνησαν, κατηγόρησαν, πρόβλεψαν μέτρα ε, για να βεβαιωθούν ότι δεν θα ξανασυμβεί κάτι ανάλογο. Αυτό συμβαίνει, το ίδιο θα συμβεί και με το περίπτωση του κ. Κασόντζη. Τη δεκαετία του 90 Ο πρόεδρο Ρίγκαν ήθελε να λύσει το πρόβλημα με το Ιράν τότε με την ανάλογη υπόθεση. Τι συνέβη. Οι ανακριτέ έλαβαν ανάλογα μέτρα ώστε να μην συμβεί κάτι ανάλογο. Ε, κατά τα άλλα, το τι συμβαίνει ακριβώ στη χώρα μα δεν είναι δουλειά σα. Είναι ένα θέμα το οποίο το αντιμετωπίζουμε. Μα πονάει μεν. Αλλά η τιμιγορία του ανώτατου δικαστηρίου έχει εκδοθεί, θα ασκηθεί έφεση και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η νομική διαδικασία. Για τον Τζαμάλ Καχρότζη. Για τους άλλους κρατουμένους, όπως είπα, με όλο το σεβασμό, δεν δεχόμαστε κηρύγματα και διδάγματα. Είμαστε ε, ανεξάρτητη χώρα. Έχουμε το δικό μας νομικό σύστημα. Θα ακολουθούμε τους δικούς μας νόμους και αυτό ακριβώ θα συμβαίνει. Εμεί δεν σα δίνουμε μαθήματα για του δικού σα νόμου και την νομοθεσία σα, ούτε για το πώ συμπεριφέρεστε στι μειονότητε. Δεν σα λέμε τι κάνατε στο παρελθόν, ακόμη και στη δική μα την περιοχή. Είμαστε κυρίε χώρε, είμαστε σύμμαχοι και είμαστε φίλοι. Υποτίθεται ότι συμβαδίζουμε σε σημαντικά ζητήματα. Αλλά δεν μπορείτε να κάθεστε εδώ και να μα δίνετε μαθήματα σε μια χώρα που είναι εθνικά απολύτω κυρίαρχη για θέματα ε, που βασίζονται σε ελλειπείς πληροφορίες και πληροφόρηση δεν είναι θεμητό, δεν είναι δίκαιο και δεν είναι και σωστό όταν μιλάτε με φίλους. Τα κάλυψα όλα. Όσον αφορά τις σχέσεις με την Τουρκία ίσως. η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα, σημαντική χώρα στην περιοχή και έχουμε εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία. Έχουμε κάποια θέματα με την Τουρκία για την ανάμειξή της στη Συρία και για το τι κάνει στη Λιβύη και προσπαθούμε να φροντίσουμε οι σχέσεις να παραμείνουν και η Τουρκία να είναι ένας υπεύθυνο παίκτη στην περιοχή που θα βοηθάει στη σταθερότητα. Πρόεδρος, αγαπητοί συνάδελφοι, πριν ευχαριστήσω τον φιλοξενούμενό μας